Ε, ομόφωνα δεκτό το ψήφισμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρακτικά θα είναι στη διάθεσή σας στην αρχή της επόμενης ε, συνόδου της Ολομέλειας. Ε, οπότε θα μεταβάσω στους αρμοδίους τα ψηφίσματα, δεν βλέπω καμία αντίρρηση και άρα διακόπτεται η Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλό ταξίδι. Λύεται η συνεδρίαση.